Κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε και βεβαρημένη μερίσια διάταξη. περάσουμε κατευθείαν στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, αν έχετε παρατηρήσεις, δεν έχετε. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. 15 ε, γλώσσες ε, είναι σήμερα το γλυσκό μας καθεστώς και περνάμε στο 3. μαθαίνουμε τις εμπορικές πρακτικές. Κύριος Ντές, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα σήμερα όπως συχνά και προηγουμένως κατά το παρελθόν. Πριν δύο ώρες πήρα τη λίστα ψηφοφοριών. Δεν μπορώ να ψηφίσω για τις αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές. Πρέπει για την επόμενη εβδομάδα να αναβληθεί η ψηφοφορία στις Βρυξέλλες για να μπορέσουμε να μελετήσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Πραγματικά ε, δεν γίνεται να λειτουργούμε έτσι. Το έχω πει, έχω ασκήσει κριτικές και θα το ξαναζητήσω. Ζητώ αναβολή για την, για την επόμενη εβδομάδα. E, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Είναι πολύ μεβαρημένη μέσα διάταξη. Αν θέλουμε να εγκριθεί αυτό το έγγραφο, κάτι από τώρα πρέπει να γίνει για να εγκριθεί σε αυτή την ε, θητεία. Δεν ξέρω, Η εισηγητής μάλλον θα μας τα εξηγήσει καλύτερα. Ή η εισηγήτρια. Κυρία Μαγκίνες. Θα λάβει πρώτα το λόγο κυρία Μαγκίνες και μετά ο κύριος Δεκάστρο. you, Chair. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στηρίζω αυτό που είπε ο Άλμπερτ και κάθε Δευτέρα απόγευμα στο Στρασβούργο είναι μια δύσκολη μέρα και εγώ έχω το Προεδρείο και άλλε ανηλυμένε υποχρεώσει. Όπω όμω σα εξηγήσει και ο συγητής, έχουμε θέματα χρονοδιαγράμματο ε, που καθιστούν λεπτό αυτό το θέμα και οι συνεργάτε μα έχουν εργαστεί νυχθημερών και στο Σαββατοκύριακο για να προετοιμάσουν ε, τη λίστα ψηφοφορίας. Στον Άλφο Άλμπερντε, που σωστά τα λέει, είναι έγκυρο το επιχείρημά του. Πρέπει όμω να καταλάβουμε ότι αν καθυστερήσουμε αυτή την ψηφοφορία, κάποιοι θα χαρούν. Όσοι δηλαδή δεν θέλουν να δουν να περάσει η νομοθεσία αυτή. Δεν ξέρω, καλύτερα να μα δώσει μια αναλυτική εξήγηση και ο εισηγητή. Ε, ναι. Εντάξει. Συμφωνώ κι εγώ. Ο κύριος Ντέ θέλει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τη δίκηση. Μία ερώτηση. Τόσο πρόβλημα είναι μία εβδομάδα για να φοβούμαστε ότι δεν θα εγκριθεί αυτή η νομοθεσία. Πόσο θα καθυστερήσουμε εάν ε, αναβάλουμε για μία εβδομάδα την ε, ψηφοφορία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι δυνατή αυτή η αναβολή. Ja myślę, że ο κ. Δεκάστρο τώρα έχει το λόγο. Και αν χρειαστεί εκπρόσωπο τη διοίκηση. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι η δουλειά που έχει γίνει Ναι, δουλεύει το μικρόφωνο μου. Ναι, μάλιστα. Ξαναρχίζω. Λοιπόν, έλεγα ότι συμφωνώ πως ε, η εργασία που έχει γίνει μας υποχρεώνει σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια και προθεσμίες. Από την άλλη πλευρά, μαζί με τον κύριο ε, όταν κάναμε το κανονισμό Omnibus για να καταφέρουμε να εγκρίνουμε έναν κανονισμό, να, φτιάξουμε τους, να, να, κάνουμε τους απαραίτητους ε, ε, τριμερείς και μαζί να ολοκληρώσουμε την εξέταση του θέματος εντός της ΙΤΕΣ, χρειάστηκε να δεχτούμε προθεσμίες πάρα πολύ στενές που μας υποχρεώνουν να ξεκινήσουμε τους τριμερείς για την οδηγία ταυτόχρονα με την ψηφοφορία στο Ολομέλεια που θα γίνει την επόμενη σύνοδο του Οκτωβρίου. Δηλαδή, Δηλαδή αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν το κάναμε επειδή μα άρεσε, αλλά επειδή ήταν η μοναδική δυνατότητα που είχαμε εάν θέλαμε να φτάσουμε σε συμβιβαστική με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ε, πριν τα Χριστούγεννα ή μάλλον μέχρι τα Χριστούγεννα. σαφώ εάν υπάρξει πολιτική συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα, εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, δεν θα έχουμε και έγκριση αυτή τη νομοθεσία μέσα σε αυτή τη θητεία. Δεδομένε τη δουλειά που κάναμε με τις συμβιβαστικέ, με το ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συνένεση για όλες τις 42 ε, συμβιβαστικέ και τις 30 για τα άρθρα και ε, τις 12 για τα εισαιτιολογικέ σκέψει ε, και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω του τεχνικούς και όλο το επιτελείο της γραμματεία για αυτό το μέγα επίτευγμα. Εάν λοιπόν δεν εκμεταλλευτούμε αυτό το παράθυρο ευκαιρία, ε, θα ε, θέσουμε ένα αμφιβόλο όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματά σας, αλλά Πραγματικά θα ήθελα να σας ζητήσω από όλους να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα για να μην διακινδυνεύσουμε να τα α, γκρεμίσουμε όλα. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά που ο κύριος Δεκάστρο, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία, παρακαλώ. Ναι, σημειώνουμε αυτό που έχετε πει. Ο Άλμπερτ όμως συνεχίζει να παραπονείται. Κύριος Άγνη τώρα έχει το λόγο. Συγγνώμη, αυτή είναι μια πολύ καινούργια. Συγγνώμη, αυτή είναι πολύ καινούργια κάρτα ψηφοφορίας, αλλά δεν δουλεύει. Μπορεί κάτι να γίνει, παρακαλώ, πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Πριν μια ώρα την πήρα, αλλά δεν λειτουργεί στο μηχάνημα. Πρόεδρος, θα ζητήσουμε τεχνική υποστήριξη θα έρθει κάποιος να σας βοηθήσει. Οπότε νομίζω τα ξεκαθαρίσαμε όλα κύριε Άγνιου. Από ό,τι φαίνεται όλα πάνε καλά τώρα. Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Δεν ξέρω να Θέλει να πει κάτι ο ή να προχωρήσουμε. Έχουμε τροπολογίες. Ε, εδώ διάφορες είναι σημαντικό το θέμα. Είπε και τα περί χρονοδιαγράμματος ε, ο κύριος Κάστρο. Έχουμε ε, την Ολομέλεια του Οκτωβρίου τη δεύτερη που θέλουμε να ψηφίσουμε. Είναι προτεραιότητα και για την Προεδρία. Ζητώ την κατανόησή σας. Λοιπόν, 61, ποιο ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. 61. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελέγχουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Πρώτο μπλοκ ή 6 συμβιβαστική άρχεται ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 6. Πρώτο μπλοκ. Πέρας ψηφοφορίας. Έγινε δεκτή η συμβαστική 6. 182. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 180. Ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 179. Α, θέλετε να ελέγξουμε την 180, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 179 ψήφι πέρι Κατά. Απορρίπτεται. 186 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Ηλεκτρονικά μάλλον ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. και τρία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με τον κύριο Αντεκάστρο πηγαίνουμε στην ΕΝΒ Ψήφι περ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ να ψηφίσουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.51 ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 2.79 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη συμβαστική 7 εγκρίνεται συν μία του εισηγητή 300 υπέρ της τροπολογίας 300 εγκρίνεται. ...297 υπέρ κατά απορρίπτεται. 299 υπέρ κατά απορρίπτεται. 21, συμβιβαστική 21, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 22. Άρχεται. Πέρας. Περνάμε στην 323. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 327 υπέρ κατά απορρίπτεται. 328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 330 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 331 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 23 άρχεται. Ο πρόεδρος μιλάει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί διαφορετικά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλες τις ψηφοφορίες. Τέλος ψηφοφορίας. Συν ένας εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την ΔΕΒΕ 13 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 224, ε, μάλλον 24 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος πληροφορίας. Εγκρίνεται. 352. Παρακαλώ. Ίσως να υπάρχει ένα πρόβλημα ο διερμηνίας. Εγώ πάντως δεν άκουσα για τη συμβιβαστική 23 τι έγινε και ούτε είδα στην οθόνη τι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Έγινε δεκτή, σας ευχαριστώ που μας το επισημάνατε. 352 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 446 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 407 υπέρ. Εγκρίνεται. Τι θέλετε. Ελέγχουμε την 407. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται. Ευχαριστώ που ζητήσατε να γίνει λεγχθή. 357 υπέρ. Εγκρίνεται. 353 υπέρ. Εγκρίνεται. 354 υπέρ. Εγκρίνεται. 358 υπέρ. Εγκρίνεται. 359 υπέρ. Εγκρίνεται. 501 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 501. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τα υπέρ. Κατά.

361 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Άρχεται η ψηφοφορία. 25. λίγη η ψηφοφορία. 29. Εγκρίνεται. 29 συμβιβαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Πέρασε. Εγκρίνεται. 384 υπέρ. Εγκρίνεται. 389 υπέρ. Εγκρίνεται. 390 υπέρ. Εγκρίνεται. Κύριε Καπούτο, να σηκώνετε το χέρι σας παρακαλώ. Δεν σας βλέπω, είστε και συντονιστής. 3,92 υπέρ. Εγκρίνεται. 3,90 υπέρ και λοιπές. Εγκρίνονται. Τις ψηφίσαμε αυτές. Πάμε στα 404 υπέρ. Εγκρίνεται. 405 υπέρ απορρίπτεται. 406 πέρ κατά απορρίπτεται. 435 πέρ. Ελέγχουμε. Την 406. Πέρασε. Odrzucona. Ε, Poprawka 435. Pani poseł Petir. jest... 435. κατά, Απορρίπτεται. 409 υπέρ. Εγκρίνεται. 412 και 14. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 413 υπέρ, εγκρίνεται. 420 και λοιπές. Υπέρ, κατά. Ε, ελέγχουμε. 4, 20, 87, 88, 33 κτλ. Υπέρ. Zamykam głosowanie. Πέρας ψηφοφορίες. Παύκα 399, Εγκρίνεται. 399 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβεβαστική 27, αρχεται ψηφοφορία. Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε. Στην 4.15 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4.16 υπέρ. Εγκρίνεται. 4.17 υπέρ. Α, να ελέγξουμε 416. Εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία. Σουβάνι 416. Πέρασε. Απορρίφθηκε με μία ψήφο 417 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 418 υπέρ. Εγκρίνεται. 422 υπέρ. Εγκρίνεται. 424 υπέρ. Εγκρίνεται. 445 υπέρ. Εγκρίνεται. 426 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 427 υπέρ, εγκρίνεται. 428 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 448 υπέρ, εγκρίνεται. 430 υπέρ, εγκρίνεται. 431 υπέρ, εγκρίνεται. 449 υπέρ, εγκρίνεται. 432 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 433 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μα καταψήφισε. Τέλο πάντων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 4-3-4 υπέρ. Εγκρίνεται. 4-5-1 υπέρ. Κατά. απορριπτηκε 4 4-3-6 υπέρ. Εγκρίνεται. 4-5-3 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε την 453. Εντάξει. Να πάω πιο πίσω θέλετε. Στην 451 θέλετε να πάμε. Εντάξει, ελέγχουμε την 451. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 436 για να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 453 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 437 υπέρ, εγκρίνεται. θέλετε να ελέγξουμε την 437, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. odrzucona jednym głosem. Απορρίφθηκε. 438 υπέρ, κατά. Απορρίφθηκε. 439. 439 υπέρ. Εγκρίνεται. 440 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Την 440. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 442 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 443. Περ. Κατά. Ελέγχουμε την 443. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 454 εγκρίνεται. 411. Υπορρίφθηκε. 354 εγκρίθηκε. Συμβαστική 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Θέλετε να ελέγξουμε κάτι. Την 454. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 28, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 470. Υπέρ. 471. 4,75 υπέρ κατά απορρίπτεται. 4,76 υπέρ κατά απορρίπτεται. 4,77 υπέρ κατά απορρίπτεται. 4,78 υπέρ εγκρίνεται. 4,79 υπέρ κατά ελέγχουμε την 4,79 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 480 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 482 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 484 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 488. Ελέγχουμε την 484. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίφθηκε. Τώρα 488 υπέρ. Εγκρίθηκε. 490 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 492 υπέρ. Ελέγχουμε τη 490 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ναι, μα θέλετε να ελέγξω. 492. Υπέρ, κατά. Κυρίες και κύριοι, μην μιλάτε. Σταματήστε να μιλάτε και σηκώνετε τα χέρια. Επαναλαμβάνω. 492. Υπέρ, κατά. Απορρίφθηκε. 496 υπέρ, κατά. Απορρίφθηκε. 497 υπέρ, κατά. ποχές, απορρίφθηκε. 498 υπέρ, κατά. Εγκρίθηκε. 500 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Άρχεται ψηφοφορία. Zamykam μου Πέρας. Περνάμε στην 508. Α, εγκρίθηκε. Πάμε, ε, πάμε στην 509, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 41, υπέρ, εγκρίνεται. 511, υπέρ, κατά απορρίπτεται 42 υπέρ εγκρίνεται 512 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 43 υπέρ εγκρίνεται 515 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 516 συν NV59 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ε, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 524 υπέρ της κυρίας Ένωρα. Κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Περνάμε στην 532. 532 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Συμβιβαστική 10, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική... <clears throat> Δεν ξέρουμε γιατί έσβησε το μικρόφωνο. 583 εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική 10 λέει τώρα ο πρόεδρος. Όχι, διορθώνουμε σε συμβιβαστική 11. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλο. Τέλος. Przyjęty. Przechodzimy do kompromisu 12. Otwieram głosowanie. Εγκρίνεται συμβαστική 12. Άρχεται. Τέλος, εγκρίνεται. 577 υπέρ, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 24 υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική 16, άρχεται. Συμβαστική 13. Τέλος ψηφοφορίας. ακριβήθηκε. Συμβαστική 14. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 595. Πετήρ υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην 599. Υπέρ. Εγκρίνεται. 600. Υπέρ εγκρίνεται. 601 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 602 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συγγνώμη, συμβαστική 15. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την συμβαστική 15. Τέλος τώρα. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 614 υπέρ. Εγκρίνεται. 615 υπέρ. Εγκρίνεται. 617 υπέρ. Εγκρίνεται. 618 υπέρ. Εγκρίνεται. 619 υπέρ. Εγκρίνεται. 620 υπέρ. Εγκρίνεται. 622 υπέρ. Εγκρίνεται. 6.24 υπέρ κατά απορρίπτεται 6.25 υπέρ κατά απορρίπτεται 6.27 υπέρ εγκρίνεται τώρα ψηφίζουμε unblock η τροπολογία για την ε, επιβολή του δικτύου σε ολόκληρη την Ένωση. Ψηφίζουμε λοιπόν unblock. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. Περνάμε στην τροπολογία DV26. DV26 υπέρ. Έκρινεται. Συμβιβαστική 18. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 18. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε να ψηφίσουμε την 48 ΙΜΚΟ. Και του κυρίου Νταντέ, υπέρ. Εγκρίνεται. 655 υπέρ. Εγκρίνεται. 657 υπέρ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Συμβαστική 19, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εκρίνεται. Περνάμε στη ψηφοφορία για τη συμβαστική 20. Άρχεται. Τέλος. Συμβαστική 20 λοιπόν είπαμε, έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 670. Υπέρ. Εγκρίνεται. 672 και 73 υπέρ κατά απορρίπτεται. 671, 674 από κοινού ε, υπέρ κατά απορρίπτονται. 675 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 676 υπέρ κατά απορρίπτεται. 677 έχει αποσυρθεί. 678 υπέρ εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία Ένα των ε, αιτιολογικών σκέψεων υπέρ εγκρίνεται. 2 το εισηγητή υπέρ εγκρίνεται. Ήμκο 1 και NV1 που είναι ταυτόσημες υπέρ εγκρίνεται. 3, 64 και 65 υπέρ εγκρίνεται 66 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ε, περνάμε στη συμβιβαστική 31 η έρτος, η 74 έρτος, έχει αποσυρθεί. Συμβεβαστική 31 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας ε, ε, εγκρίνεται ε, τροπολογία 77 Αγγιλέρα. Υπέρ εγκρίνεται MV3. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Υμκο, 4. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32 άρχεται. Εγκρίνεται η συμβιβαστική και πάμε στην 89 Νταντά. Και λέω και το όνομα για να βρείτε ποια τροπολογία είναι. Υπέρ, ε, εγκρίνεται. 8 του εισηγητή και ΙΜΚΟ. Ε, υπέρ ποιοι είναι, εγκρίνεται. Τροπολογία 90, υπέρ, κατά, <clears throat> απορρίπτεται. 91, υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Οτιέρα, <clears throat> Odrzucona. Poprawka... Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ήμκο. Ε, υπέρ εγκρίνεται. 92. Υπέρ κατά ε, απορρίπτεται. 93. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Δεύε 5. Υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική 33. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34. Άρχεται. 34 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 116. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 35. Άρχεται. εγκρίνεται. Συμβαστική 36 άρχεται. Τέλος, εγκρίνεται. Συμβαστική 37 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Συμβαστική εγκρίνεται. Συμβαστική 38 άρχεται. <coughs> Τέλος. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά απορρίπτεται. 136 υπέρ εγκρίνεται. 138 υπέρ εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Για μία ψήφο. Τροπολογία 141. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 142. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 39. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 154. Ζα. Υπέρ κατά, υπέρ Συμβαστική 40 ψηφίζουμε. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40, συμβιβαστική 41. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική 42. <coughs> Εγκρίνεται και περνάμε σε 170. Νταντά, υπέρ, εγκρίνεται. 19 το εισηγητή, υπέρ, εγκρίνεται. Ήμκο, υπέρ, εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες, δες, γιάρ, έρτος, ένρα, υπέρ, εγκρίνονται. 174. Ε, συγγνώμη, 178 υπέρ κατά απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Ποιο είναι το πρόβλημα?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 already of these amendments, but we went immediately to CA4. This amendment. Yeah, yeah, but first we have to see what happened to NV18. Głosujemy jeszcze raz, głosujemy nad poprawką. Och, ξαναψηφίζουμε την τροπολογία NV18 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. NV18. Σελίδα 4 λέει ο πρόεδρος, εμείς δεν έχουμε καμία σελίδα εδώ. NV18. Ψηφίζουμε για την NV18. Τέλος. Ένας παραπάνω FDD, η FDD ψήφισε. Τέλος ψηφοφορίας. Πρόεδρε, τρεις. Τρεις είναι οι FDD εδώ και έχουν και τρεις ψήφους. Ναι, δίκιο έχετε, αλλά αυτό το μηχάνημα δείχνει πως είναι ένα παραπάνω, παραπανήσιος διευθυντή. Μα μην εμπιστεύεστε τα μηχανήματα, ποτέ. Ναι, ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τέλος της ψηφοφορίας απορρίφθηκε Η τροπολογία 2.42, αν κατάλαβα καλά, την ξεχάσαμε. Υπέρ. Rejected, yes, 39. 242, 240, 242 και στη συνέχεια έχει μερικές Następnie... 39 και τα λοιπά. σελίδα, τέσσερα είμαστε πάντα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. «246-248. Μαγκίνες. Να ψηφίσουμε και τη 250. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ε, Τελική ψηφοφορία τώρα για την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Με ονομαστική κλίση άρχεται. Τσιέραμ, Ζαμεκάμ. Τέλος. Εγκρίθηκε. σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται. Zagłosowali Państwo? Tak, Ψηφίσατε όλοι, μάλιστα. Τέλος ψηφοφορίας. Okay. Εγκρίθηκε. Περνάμε και στην επόμενη σε ψηφοφορία για να προβούμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σύμφωνα με το 32, άρθρο 32 και για τη σύσταση της διαπραγματεύτική ομάδας άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Ε, να μην δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Το αξίζει, συγχαρητήρια. Ναι, να σας να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά όλους τους συναδέλφους ε, τους ε, σκιώδεις Μαγκίνες, ε, μακιντάρ, Κατάινεν, Κάρθη, Μαρία, Σούλα. <clears throat> Όλοι δούλεψαν πάρα πολύ, γι' αυτό και πετύχαμε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία. Θα μπορέσουμε έτσι νομίζω να φτάσουμε, ελπίζω, ελπίζω, ναι όλους τους σκιώδες να τους ευχαριστήσω. Θα φτάσουμε λοιπόν πολύ ισχυροί στην Ολομέλεια στις 22. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το τεχνικό μας επιτελείο που δούλεψε νυχθημερών και ταυτόχρονα βέβαια και την γραμματεία Βασίλη όλους σας. Σπουδαία δουλειά και βεβαίως τώρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε θα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε εντός της Αυστριακής Προεδρίας. Panie Σας ευχαριστούμε και εμείς αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Και εμείς έχουμε πολλή δουλειά και οι συνεργάτες μας. Η γραμματεία, οι σκιώδης. Πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ καλό να ολοκληρώναμε αυτό το θέμα εντός της ε, θητείας αυτής γιατί έτσι θα στείλουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Ε, είχαμε την έκθεση ΙΜΚΟ, Μαγκίνες, ανέλαβε την ευθύνη της έκθεσης, προχωρήσαμε, μετά είχαμε μία σύγκρουση μεταξύ των επιτροπών. Τουλάχιστον ε, μπορέσαμε και ψηφίσαμε σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό και είναι σημαντική η συμβολή. Εγώ σημείωσα βέβαια αυτά που είπε ο κύριος ε, Ντές ε, και ε, για τον κύριο Καλινός. Τέλος πάντων, τι να κάναμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώ. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε με το, στο σημείο 4 της ε, διάταξη. Ε, διάταξης. Κύριε Καλινός, και ναι, πράγματι πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, για τη αντίκτυπο ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον εισηγητής είναι ο κύριος Ροπέ. Αν θέλετε σύντομα παρακαλώ για να σας δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλή πρόταση της Επιτροπής, φιλόδοξη. Συνεργάστηκα πολύ καλά με τους κοιόδης και τη γραμματεία. Χαίρομαι γιατί όλοι συμμετείχαν ενεργά. Είχαμε 215 τροπολογίες, δεν και λίγες. Δεν ήμασταν καθήλια αρμόδια επιτροπή. Γνωμοδότηση συντάξαμε Envy είναι η αρμόδια. Η Envy είναι αυτή που θα λάβει την τελική απόφαση. Θέλαμε όμως να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλαμε να εστιάσουμε στα πλαστικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Γιατί η πρόταση της Κομισιόν δεν ήταν επαρκής ως προς αυτό το σημείο. Τα πλαστικά απορρίμματα μολύνουν τις θάλασσες και τα ύδατα αλλά και τα μικροπλαστικά είναι ένα θέμα που θέλαμε να αναφέρουμε και θέλαμε να δώσουμε έμφαση στο ότι είναι διαφορετική η κατάσταση με τα μικροπλαστικά ανάλογα με την τοποθεσία, με το μέρος. Ε, υπάρχουν ε, μέρη στα οποία μπορεί να αποσυντηθεί πάρα πολύ εύκολα, το μικροπλαστικό σε άλλες όχι, τέλος πάντων. Πρόεδρος, ναι, πράγματι είναι σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα για τα μικροπλαστικά ούτε καν ήξερα πόσο σημασία έχουν αυτές οι πτυχές. Να περάσουμε όμως τώρα στην ψηφοφορία παρακαλώ τη συνάδελφοι. ...94 υπέρ, εγκρίνεται. 96 Περ. Εγκρίνεται. 98 υπέρ, εγκρίνεται. 99 υπέρ, εγκρίνεται. 106. 106. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. 100. Ε, Ελέγχουμε. Την 105. Πέρας. 107, Κατά, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβιβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, 9 διορθώνει ο πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 176. 176 καπούτο υπέρ Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Έχουν γίνει δεκτές όμως οι συμβιβαστικές, οπότε πηγαίνουμε στη σελίδα 9. Συμβιβαστική 0. Σελίδα 9. Έτσι λέει τουλάχιστον το δικό μου το χαρτί, γιατί έχουμε ψηφίσει όλες τις προηγούμενες συμβαστικές, πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή και συμβιβαστική 0. Πηγαίνουμε τώρα στο τροπολό 29 Χάζεκαμπ. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Σε σκέψεις πάμε τώρα. 5 και 5 Αλφα. Όχι, ελέγχουμε την τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 29 τροπολογία. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τώρα λοιπόν τελικέ σκέψεις. Α, όχι. Όχι, πάμε στην τροπολογία 40. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 40. Κατά, ποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Άρχεται ψηφοφορία. Αν γίνει δεκτή, η 40 Έρχομαστε στην συμβαστική 2. Εδώ είμαστε τώρα, ψηφίζουμε, συμβαστική 2. Είχε απορριφθεί όμω ε, η 40, άρα πρέπει να ψηφίσουμε τη 41. Ποιο είναι υπέρ τη 41, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο, συγγνώμη. Απορρίφθηκε. Τώρα πηγαίνουμε συμβαστική 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 53. Νταντά. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 53. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 56. Όχι, 55 πρώτα, διορθώνει ο πρόεδρος ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. Τώρα 56 υπέρ. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 59. Άρχεται η ψηφοφορία. 59. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 63 υπέρ. Εγκρίθηκε. 64 υπέρ. Εγκρίθηκε. 65 υπέρ. Εγκρίθηκε. 66 υπέρ. Εγκρίθηκε. 67 υπέρ της 67 κατά ελέγχουμε την 67 άρχεται η ψηφοφορία 67 πέρας απορρίφθηκε 68 υπέρ κατά απορρίφθηκε 69 υπέρ εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Υπέρυπα. Κατά απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 77 υπέρ, εγκρίνεται. 78 υπέρ, εγκρίνεται. 79 υπέρ, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 8. Το εισήγητη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Εγκρίνεται. 84. 84 υπέρ. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. απορρίπτεται. 85 υπέρ, εγκρίνεται. 86 υπέρ, εγκρίνεται. 87 υπέρ, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 10 εγκρίνεται. Άρχεται λοιπόν τώρα η ψηφοφορία του συνόλου της έκθεσης. Εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότηση. συγχαίρουμε και τον εισηγητή. Θέλετε μήπως το λόγο? Αν όχι, τότε περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, την έκθεση Μπούντα. Ναι, έχετε το λόγο. Τα ξέρετε καλύτερα να μας τα πείτε. Ναι, σα ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το λόγο έχει ο κύριο Καπούτο, γιατί αυτού είναι η έκθεση τώρα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα πάτε πάρα πολύ γρήγορα και <clears throat> με πιάσατε απροετοίμαστο. Λοιπόν, είναι μια τεχνική τώρα γνωμοδότηση που έχει ε, παραλείπτει την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Πολλές τροπολογίες στόχο έχουν να αυξήσουν τη διαφάνεια προς τους ε, πολίτες και να απλοποιήσουν την επικοινωνία ώστε να βελτιωθεί λοιπόν η επικοινωνία και η παρακολούθηση της εφαρμογής ε, της οδηγίας για το περιβάλλον. Δεν υπήρξε, υπάρχει, υπήρξε λόγος να κάνουμε συμβιβαστικές γιατί όπως σας είπα είναι μια απλή τεχνική έκθεση, οπότε απλά πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. E, ναι, είναι δύσκολο να υποβάλει κανείς εδώ συμβιβαστικέ τροπολογίες, οπότε ναι, θα περάσουμε στην τροπολογία. 4 καπούτο υπέρ. Εκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 10 υπέρ κατά απορρίπτεται 11 υπέρ κατά απορρίπτεται 12 υπέρ κατά απορρίπτεται 13 <clears throat> υπέρ κα, εγκρίνεται περνάμε στα 15 καπούτο υπέρ εγκρίνεται 16 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 16. Zamykam głosowanie. Τέλος. Απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ε, 19 υπέρ εγκρίνεται. 20 υπέρ εγκρίνεται. 21 μέχρι και 23 καπούτο υπέρ κρίνονται 24 υπέρ κατά απορρίπτεται 25 υπέρ κατά απορρίπτεται 26 υπέρ κατά απορρίπτεται 27 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27 Απορρίφθηκε. 28 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 31 υπέρ, α, συγγνώμη, εγκρίθηκε. 31 υπέρ, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 33. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 34 λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. Εγκρίθηκε. Προπολογία 35 υπέρ κατά επαληθεύουμε έρχεται τέλος απορρίφθηκε 36 υπέρ κατά απορρίπτεται 37 υπέρ κατά επαληθεύση τέλος εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 ε, υπέρ εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά για τη 40. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Gdzie my jesteśmy? 40. Poprawka 40. Kto... 40 υπέρ. Όχι, την κάναμε. 41-42 από κοινού, unblock. Ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ Η πρώτη έχει καταπέσει. Δεύτερη παράγραφο τη 43. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Τροπολογία, ε, παράγραφος 2 λοιπόν, 43-2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, εγκρίνεται. 44, υπέρ, κατά, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Φιέρα πληροφορία. Ζαμίκα. Τέλος της πληροφορίας απορρίφθηκε η τροπολογία 45 τώρα υπέρ κατά απορρίπτεται 46 υπέρ εγκρίνεται 47 υπέρ εγκρίνεται 5 υπέρ εγκρίνεται 6 υπέρ εγκρίνεται 7 υπέρ εγκρίνεται 1 καπούτο εγκρίνεται Ψηφίζουμε για το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική κλίση. Τέλος. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Και Καπούτο, θέλετε το λόγο? Όχι. Ωραία. Περνάμε λοιπόν την έκθεση του κυρίου Μπούντα, στον οποίο δίνω το λόγο. Δεν έχω κάποια παρέμβαση. Είναι πολύ σαφής η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε. poprawki pierwsza i druga odrzucające propozycję komisji. E, kto jest Ποιο είναι υπέρ τη πρόταση Κομισιόν. Α, όχι. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. όλοι ήταν υπέρ. Όμως πρέπει να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση. Γιατί έχουμε και κάποιες τροπολογίες. Να ξαναψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Ο Φίλιπ να μας ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα θέλει τώρα. Νομίζω είναι σαφής η ιστορία. Οι τροπολογίες για την απόρριψη της ε, πρότασης έχουν εγκριθεί ομόφωνα και τώρα ψηφίζουμε για να εγκρίνουμε την γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Αν είστε υπέρ της απόρριψης θα πρέπει να ψηφίσετε ναι. Θα πρέπει να ψηφίσετε υπέρ. Για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση δεν ψηφίζεται επί της πρότασης, αλλά επί της γνωμοδότησης που απορρίπτει την πρόταση. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν, η τελική ψηφοφορία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 Μέσα σε μια ώρα και δέκα λεπτά τα ψηφίσαμε όλα. Ήμασταν πολύ γρήγοροι. Χάρη στον κύριο Καλινόσκι. Α, και σηκώθηκε να φύγει. Και αυτό βιαζόταν. Τώρα το κατάλαβα. Żyje. To? το poseł Kalinowski και μου έδωσε ένα ωραίο νέο που δεν θα σας το μεταφέρω όμως. Για το θέμα τα είναι εδώ ο εισηγητής. Ο κύριος Ματ Κάρθη. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις Βρυξέλλες, ε, για την επίσκεψη, αλλά εδώ είναι ο κύριος Κάρθη και θέλει το λόγο νομίζω. όκ. Ε, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία. Είχαμε κάποιες δυσκολίες για να βρούμε τον κατάλληλο χρόνο για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τα μέλη που ε, παρέμειναν τόσο αργά. Θα είμαι σύντομος όμως, όσο το δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια ο αριθμός των δασμολογικών ποσοστώσεων στον ΠΟΕ αυξήθηκαν για να αντανακλούν τις ε, αντισταθμίσεις που δίνονται στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ε, στην ε, λύση κάποιων διαφορών, εμπορικών διαφορών. Με το Brexit έχουμε την ανάγκη να κάνουμε το αντίθετο από ό,τι κάναμε στο παρελθόν, δηλαδή την επανακατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την, και, και την Μεγάλη Βρετανία. Ως μέλη θα γνωρίζουμε ότι ο γεωρικός τομέας είναι ο μοναδικός ε, που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό γιατί ο κατάλογος αυτών των δασμολογικών ποσοστώσεων είναι κυρίως ε, σε γεωργικά προϊόντα και αυτές οι ποσοστώσεις έχουν τύχη διαπραγμάτευσης με τους εταίρους που στηρίζονται σε ευαίσθητες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις της αγοράς να απορροφήσει τα αγαθά και να διατηρεί τιμές για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Άρα για την επανακατανομή αυτών των ποσοστώσεων και η μεθοδολογία θα πρέπει να αναγνωρίζει την ευπάθεια κάποιων τομέων και την πιθανότητα αυτών που ε, παράγονται σε διάφορες αγορές. Ε, η μεθοδολογία είναι κάτι η οποία έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στους εταίρους. Πρέπει να διασφαλίζει μια δίκαιη κατανομή των παραχωρήσεων ανάλογα με το μερίδιο χρήση του κάθε εταίρου, άρα δεν προτείνω ε, τροπολογίες σε αυτό, αλλά αυτό που μόνο του δεν διασφαλίζει ε, μια δίκαιη και ισορροπημένη ισορροπία των ΔΠ, γιατί μπορεί να ε, τροποποιηθούν αυτοί οι αριθμοί και σε μεταγενέστερο στάδιο. Πρόεδρε, το Brexit ε, είναι καθοδόν και ε, υπάρχει ανασφάλεια σε ό,τι αφορά την τελική ημερομηνία αποχώρησης, άρα θα πρέπει να γίνουν και άλλες ε, ε τροποποιήσεις. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να έχει απεριόριστες διακριτικές ε, δυνάμεις για την επακανανομή των ΔΕΛΤΑΠΗ. Χωρί ε, την συνένεση του Ευρωκοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση, να έχει κάτι εξουσιοδότηση ε, και που έχουν γίνει συμφωνίε. Ωστόσο, για όλε τι άλλε τροπολογίε, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο σύμφωνα με τι ε, διαδικασίε. Σω να φαίνεται τεχνική αυτή η άσκηση, και επειδή δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη λύση για να ε, αποφευθεί το δυσπροπέλαστο σύνορο με την Ιρλανδία. Συμφώνησαν ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Έννοία αγορά και την Τελεωνιακή Ένωση. Αυτή οι, αυτές οι θα, πρέπει να οδηγήσουν σε άλλη επανακατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων. Και αυτό θα υπέχει, ε, υπέχει πολιτικές αποφάσεις. Επίσης, όπου υπάρχουν, όπου το μερίδιο χρήσης των Βρετανικών ποσοστώσεων είναι χαμηλό, τότε ε, ίσως ε, να οδηγήσει σε μικρότερο ποσοστό, ε, άρα θα μπορεί να χρειάζεται διαφορετική αποστολή, ε, θα πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση και πρέπει αυτό να περάσει από κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ε, θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατική συνένεση ε, για τις αρχικές διαπραγματεύσεις όλων των δασμολογικών ποσοστώσεων. Γι' αυτό η επανακατανομή απαιτεί την ίδια επίβλεψη. Δουλεύουμε με στενά χρονοδιαγράμματα γιατί έχουμε μέχρι αύριο την προθεσμία για τις τροπολογίες. Ε, θέλουμε να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα στην Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα των δεσμολογικών ποσοστώσεων ε, γιατί όταν αυτά γίνουν λάθος, ε, τότε αυτοί που υποφέρουν είναι οι γεωργοί και οι κοινότητες που εξαρτώνται από αυτούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Πραγματικά είναι άκρος ε, σοβαρό και σημαντικό το θέμα. Θέλουμε να ονομοδοτήσουμε στην Επιτροπή Εμπορίου. Να δώσω το λόγο στους και όσοι καταρχάς. Κυρία Μίλλερ. Αξιότιμε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, γνωμοδότηση. Ουσιαστικά πρόκειται για τις δασμολογικές ε, ποσοστώσεις ε, για τα υπόλοιπα κράτη και το πώς θα ανακατενεμηθούν εντός του ΠΟΕ από εδώ και πέρα. Είναι σημαντικό πραγματικά να εργαστούμε με επιμέλεια έχοντας υπόψη μας την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου για πρέπει να προετοιμαστούμε και Πραγματικά θεωρώ ήταν πάρα πολύ καλή και επίσκεψη, όπως είπατε και εσείς, επίσκεψη στην ε, Ιρλανδία ε, δεν ε, ήξερα εγώ πραγματικά πόσο σοβαρές επιπτώσεις θα είχαν αυτά τα θέματα και τις, θα επηρέαζε τις σχέσεις Ευρωλανδίας και Ιρλανδίας. Το θέμα είναι οι κανόνες που θα ισχύουν και πραγματικά πρέπει ε, και το καταλάβαμε αυτό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα και γι' αυτό και με πολύ μεγάλη χαρά συνεργάστηκα με τον εισηγητή και εφόσον χρειαστεί θα καταθέσουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ, κυρία Σκότα. Είναι σημαντικό να ε, ε, είμαστε στο ίδιο μήκος ε, και είμαστε κυρία Σκότ κάτω. και σίγουρα μας βρίσκει σύμφωνο σε ανάγκη τήρησης των κανόνων του ΠΟΕ. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, διαφάνεια αν χρειαστεί προσαρμογές στον κανονισμό. Επειδή όμως ε, γίνεται ένας χαμός ε, με το Brexit και με τα όσα προτείνει ο Τραμπ που διαταράσει την παγκόσμια τάξη, ήταν ε, καλό που τον Οκτώβριο πέρυσι έγινε πολύ γρήγορα η σχετική συμφωνία, αλλά... Ίσως να είναι και αισιόδοξα τα όσα λέγονται ότι θα υπάρξει συμφωνία αποχώρησης που θα είναι η βάση για την εύλογη αυτή πρόταση. Αν υπάρξει πρόβλημα, η Κομισιόν θεωρεί ότι θα υπάρχει μια δίκαιη διαδικασία στο πλαίσιο των μηχανισμών πλήξης διαφορών του ΠΟΕ. Πριν δύο χρόνια μπορεί να ήταν αυτό μια πιθανή υπόθεση, αλλά τώρα έχουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών. Η Βρετανική κυβέρνηση υπονομεύει και την αξιοπιστία απειλώντα να αποδυναμώσει τις συμφωνίες. Άρα ποιο είναι ο έντιμος συνομιλητής ή αξιόπιστος εταίρος. Σωστά η Κομισιόν λέει ότι το Βασίλειο θα σεβαστεί τους όρους της προσωρινής συμφωνίας για τις ΔΕΛΤΑΠ. Αλλά να μην, είμαστε, να μην επαναπαυθούμε γιατί μπορεί να προκύψουν ε, καταστάσεις ε, έκτακτες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ εκπροσωπώ την ε, νοτιοδυτική Αγγλία και εδώ εκπροσωπώ πολλούς αγρότες από την περιφέρειά μου. Είναι καλή η σαφήνεια μέσω των ΔΕΛΤΑΠΗ, αλλά να μην τους δώσουμε ψευδείς ε, διαβεβαιώσεις. Και ελπίζω να μην ε, απειληθεί ούτε η νομική σχέση φύση της δραστηριότητά τους, ούτε και η επιβίωσή τους στο μέλλον. Oui, merci, euh, Τόσο χαμηλές, ε, χαμηλή τελωνιακή δεσμή δεν επιτρέπουν ε, ε, επαρκή προστασία των ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών και το να τα αφήνουμε εκτεθειμένα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι ένα μέγα σφάλμα που εξηγεί και τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί. Είναι καλό να εκμεταλλευτούμε την αποχώρηση των Βρετανών από την Ένωση για να ξεκινήσουμε πιο βαθύ προβληματισμό όσον αφορά την, την προσκόλλησή μας σε αυτή την ιδεολογία του φιλελευθερισμού που τελικά έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Δεν είναι δίκαιο να αμφισβητήσουμε το σύνολο των γεωργικών προϊόντων ε, θα πρέπει καλύτερα να προστατεύσουμε του τομεί που, που αντιμετωπίζουν σήμερα δυσκολίε. Ε, επειδή έχει αποτύχει τελείω αυτό το σύστημα ΓΚΑΤ η ε, η Κομισιόν θα πρέπει να μπορέσει να μας εγγυηθεί πως κανέναν μια ποσόστοση δεν θα αυξηθεί μετά από την ε, τέλος αυτών των διαπραγματεύσεων. Πώς θα μας το εγγυηθεί αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Νίκολσον. Κάποια πράγματα έχουν καλυφθεί, αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένε δεσμεύσει όσον αφορά του δασμού απέναντι στον ΠΟΕ. Αυτό ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέσα στην Ένωση. Το, η αποχώρηση τη Βρετανία είτε γίνεται δεν γίνει, όποτε και αν γίνει ή δεν γίνει, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να, μέχρι τότε θα πρέπει να ισχύει ε, πλήρως το σύστημα και για τη Βρετανία. Εάν δεν υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσει, ε, ε, θα πρέπει να λήξει το σχετικό καθεστώς ήδη από ε, το Μάρτιο του 2019. Διαφορετικά, το 2020 θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Σύμφωνα με τον το τελευταίο υπολογισμό τη μεθοδολογικής ανάλυσης, αυτή η μεθοδολογία βασίζεται στις ιστορικές εμπορικές ροές. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως προσπαθεί να θα πρέπει μάλλον να τηρήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις ως μέλος της Ένωσης και ως ε, αναφορά τις υποχρεώσεις για το εμπόριο και τα αγαθά. Εν γέννη υπάρχει θετική συνεργασία και έχει υπάρξει κάποια καλή πρόοδος ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη των 27. Τώρα όσον αφορά την γνωμοδότηση θα πρέπει να ζητήσω την τροπολογία 2 του εισηγητή όπου κάνει μια αναφορά που προσπαθεί να μετακινήσει το τέρμα στην μεθοδολογία την αρχική που έχει χρησιμοποιηθεί όσον αφορά τις ποσοστώσεις. Και στην τροπολογία 29 η αιτιολόγηση λέει ότι η απουσία οποιασδήποτε άλλη λύση για, για τα σύνορα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ένωση συμφώνησαν ότι η Βόρειος Ιρλανδία θα παραμείνει σε ε, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό δεν ισχύει γιατί το Δεκέμβριο του 2017 η Βρετανική κυβέρνηση και η Κομισιόν συμφώνησαν ότι η απουσία συμπεφωνημένων λύσεων ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, θα προστατευθεί η Συμφωνία του 1998 μεταξύ Βόρειας και ε, Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Αν τύχει διαφορετική μεταχείριση η Βόρεια Ιρλανδία, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε 10-20 χρόνια. Αν ισχύσουν δηλαδή διαφορετικέ νομοθεσίε ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία, δεν πρόκειται να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, άρα θα πρέπει να μα προβληματίσει. Επίση, ψευδεί ειδήσει έχουν αναπτυχθεί, ειδικά στι Βρυξέλλε, η ιδέα δηλαδή ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα είναι κομμάτι τη επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ το υπόλοιπο το Ηνωμένο Βασιλείο εκτό. Κάτι τέτοιο θα είχε πολύ σοβαρέ συνταγματικέ και δημοκρατικέ επιπτώσει για του παραγωγού στη Βόρεια Ιρλανδία. Θα είχε επίση οικονομικέ ε, επιπτώσει για του παραγωγού στη Βόρεια Ιρλανδία, γιατί σε όλου τους τομεί ε, της Γεωργίας η Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η Μαράιντε Μακίνες είναι σκιώδη εισηγήτρια για το ΕΛΚ για αυτό το θέμα. Ζητά συγγνώμη διότι δεν μπορεί να είναι σήμερα ε, μαζί μας γιατί προεδρεύει αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια. Και γι' αυτό μου ζήτησε να διαβάσω μια σύντομη δήλωση εξ ονοματός της. Λέει λοιπόν ότι θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την εργασία τους για αυτό το σημαντικό τομέα και κάνει τρεις πατρίσει. Πρώτον ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, ακολουθία, τη συνέχεια των εμπορικών σχέσεων με χώρες εκτός της Ένωσης μετά το Brexit, που θα πρέπει να συνεχιστούν ως ε, έχουν και σήμερα. Ωστόσο, δεδομένες της ευαισθησίας ε, των προϊόντων που καλύπτονται από το TRQ, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε ο κανονισμός αυτός να μην θέσει σε μειονεκτική θέση τους παραγωγούς της Ένωσης, ακόμα και χωρίς να το θέλει. Αυτέ οι διαπραγματεύσει στον ΠΟΕ δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια γενική αναδιαπραγμάτευση πρόσβαση των προϊόντων στην αγορά τη Ένωση Και κλείνει λέγοντα ότι προσβλέπει στη συνεργασία με τον εισηγητή. Σα ευχαριστώ. Oui, Monsieur le Président. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Με την γνωμοδότηση του γητού μου γεννήθηκαν κάποιε παρατηρήσει σε κάποιε συγκεκριμένε προτάσει που θα ήθελα να σα μεταφέρω. Είναι σημαντικό οι ποσοστό που χρησιμοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο των εμπορικών του με χώρε να ακυρωθούν και να μην αναδιανεμηθούν. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να επαγρυπνήσουμε για την αξιολόγηση των ε, τασμολικών προσθέσεων να δούμε πώ θα χρησιμοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο, για να μην έχουμε πλεόνασμα εξαγωγών που θα αποσταθεροποιήσει τι ζωικέ αγορέ των κρατών μελών, που είναι ευαίσθητα και βάλλοντα κλιμα, στι κλιματικέ αλλαγέ. Και θα πρέπει η Κομισιόν, κατά την άποψή μα, να έχει περιορισμένη εξουσία για να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί και να αλλάξει ε, υποφιλία τη κάποιε εμπορικέ συμφωνίε και χρειάζονται επίση έλεγχοι επικύρωσαν για τις χώρες μέλη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και κατά τα λοιπά θα στηρίξουμε τον εισηγητή στην ανάλυση του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση του έντραφου Ματ Κάρθη είναι ισορροπημένη. είναι μια καλή πρόταση. Ξέρουμε βέβαια όλοι ότι οι αγρότες μας ανησυχούν, αγωνιούν. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό που είναι στο δημοψήφισμα, γιατί αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να υπάρξει μια αναλογική μείωση των ποσοστώσεων. Οι κτηνοτρόφοι στον τομέα των προβάτων ε, στη Βουλγαρία και φαντάζομαι και σε άλλους τομείς. Παρακολουθούμε αγωνία τις εξελίξεις. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε σε άγνοια και πρέπει δίκαια να ανακατανύουμε τις ποσοστώσεις. Thank you. Ο κύριος Καπούτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφο Μακάρτη για την εξαιρετική του δουλειά γιατί εστιάζει την προσοχή σε πρακτικές επιτυχίες που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Να γνωρίζω ότι η φύση των διαπραγματεύσεων για το Brexit και τη αβεβαιότητα για την ημερομηνία και τις συγκεκριμένες συνθήκες αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να καταστήσουν ε, ε, απαραίτητες ε, τις δασμολογικές αλλαγές στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να τονιστούν άλλα στοιχεία για την νέα κατανομή, όπως ας πούμε μέτρα αγιονομικά και φυτογειονομικά για την περίοδο αναφοράς 2013-2015 που οδήγησαν σε αναταραχές, αναταράξεις με, στις συναλλαγές με συγκεκριμένο εταίρος μας στο ΠΟΕ. Αυτό σημαίνει πως ε, η ε, ότι η, δεν ε, ακολουθούμε πάντοτε τις πληροφορίες γιατί είναι ένα παράδειγμα. Είναι και οι πολιτικές αποφάσεις που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις γεωργικές αγορές που είναι πολύ ευαίσθητες κατά τη γνώμη μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει διακριτική ευκαιρία περιόριστη για να τροποποιήσει την υποδιέρεση των ποσοστό, δασμολογικών ποσοστώσεων χωρίς έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως όπως εξάλλου προτείνεται σε αυτή την έκθεση. Εγώ προτείνω πλήρη διαφάνεια και κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα έπρεπε η Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να υιοθετεί ε, εξουσιοδότηση πράξη μόνο την παρουσία μιας διεθνούς συμφωνίας γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η έγκριση από πλευρά του Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή Επιμένω η Κομισιόν να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τον κύριο Κάρθι, άκουσα και τον Τζιμ Νίκολσον και ενώ ο κύριος Κάρθη μίλησε κάτι για το οποίο ανάφερε Βόρεια Ιρλανδία, σημαίνει δηλαδή την Κομιτεία των Εγκόλ κανονικά, ενώ υπάρχει περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι η Βόρειο Ιρλανδία, είναι κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν πρόκειται να έχει διαφορετική μεταχείριση από την υπόλοιπη Βρετανία μετά το Brexit, ούτε για του δασμού ούτε και για οτιδήποτε άλλο. Ο κ. Τζιμ Νίκολσον ε, είπε ότι κυκλοφορούν διάφορε φήμε στι Βρυξέλλε ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί. Ε, και δεν το βλέπουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση. Η Βόρεια Ολλανδία είναι κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου και θα ε, έχει την ίδια μεταχείριση με την υπόλοιπη χώρα. Thank you, Chair. I should also like to thank the, the rapporteur for his draft opinion and more generally your committee for, for the interest in this file, which is indeed very technical but political. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης τα, και τους ε, σκιώδεις. Ε, αυτό καλό νέο είναι ότι έχουμε κοινό στόχο, δηλαδή την ρύθμιση των δεσμολογικών ποσοστώσεων όταν το η Βρετανία αποχωρήσει από την Ένωση. Και αυτό αποκομίζω ε, από τη σημερινή συζήτηση και από τις προηγούμενες συζητήσεις. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, χρόνος προθεσμίες. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η Κομισιόν διαπραγματεύεται με το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή που προβλέπει μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος του 2020 και αν αυτή η συμφωνία αποχώρηση ολοκληρωθεί και αρχίσει να ισχύει, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει τη Τελωνιακή Ένωση μόνο τότε. Θα έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω δηλαδή. Επίσης πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία αποχώρησης. Και άρα θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Τελωνιακή Ένωση τα τέλη Μαρτίου του επόμενου χρόνου. Και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε υποβάλει την πρόταση. Για να, να γίνουν όλα αυτά η Κομισιόν θα πρέπει να υιοθετήσει μια εφαρμοστική πράξη πολύ τεχνική φύση. Χρειάζεται λοιπόν αυτό ο κανονισμό να εγκριθεί μέχρι τα τέλη του έτου. Δυστυχώ λοιπόν βιαζόμαστε. Το δεύτερο αφορά ε, την ε, τροπολογία που είναι η βασικότερη, δηλαδή η κατάργηση του πεδίου εφαρμογή άρθρο 3. Το Συμβούλιο έχει εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες και εμείς είμαστε βεβαίως έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και με την ΙΝΤΑ αλλά και με το Συμβούλιο ώστε να βρούμε μια καλή λύση για να περιχαρακώσουμε και να ορίσουμε καλύτερα τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σε αυτό το άρθρο, ώστε να μην φαίνεται σαν να είναι απεριόριστες. Εγώ ήθελα να προτείνω να καταργήσουμε τη ρήτρα για τον ΠΟΕ θα διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας στη Γενέβη και θα πρέπει εκεί να το πείσουμε ότι οι υπολογισμοί μας γίνονται επί της καλύτερης δυνατής βάσης, ότι δηλαδή τα νούμερα είναι σωστά. Και δεν θέλουμε οι εταίροι μας να έρθουν με καλύτερα στοιχεία από αυτά που έχουμε εμείς. Γι' αυτό το και μόνο το λόγο προτείναμε αυτήν την ε, χειραφέτηση στο Β, ώστε δηλαδή να μπορέσουμε να εντάξουμε τα στοιχεία στο παράρτημα για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Αυτό για περίπτωση διευθέτησης διαφορά στην Κομισιόν και φυσικά θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο ε, πλήρως γιατί μιλάμε για τα εξουσιοδότηση πράξη θα μπορείτε να ελέγξετε και να απορρίψετε ενδεχομένω αυτό που κάνουμε αν δεν είστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμεί ευχαριστούμε. Τώρα ο εισηγητή έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες εισηγητής και όλους τους υπόλοιπου βουλευτές για την ε, συνεισφορά τους. Το χρονοδιάγραμμα σας το παρουσίασα είναι πολύ στενά τα περιθώρια και αυτό λέει πολλά και από πολλές πλευρές. Ίσως ε, να είναι το πιο εύκολο στοιχείο των διαπραγματεύσεων ε, του Brexit, γιατί έχουμε μία πρόταση από την Κομισιόν που το καταδεικνύει χωρίς μικρόφωνο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ελπίζω ότι θα έχουμε μία στερεή, αποφασιστική ε, θέση. Ως Κοινοβούλιο θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για την παρέμβασή της. Ό,τι δεν αφορά τους συναδέλφους και αυτά που είπαν για στήματα που αφορούν γειτονικέ επαρχίες ε, στη δική μου περιφέρεια για το τι θα γίνει μετά τις διαπραγματεύσεις ε, του Brexit, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ποια είναι η δική μου επιθυμία. Η δική μου επιθυμία είναι οι αγρότες στις έξι επαρχίες της ή του βορρά της Ιρλανδίας ε, ε, να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση και στη Βρετανική και στην Ασιακή αγορά και ελπίζω οι αγρότες στη δική μου την περιφέρεια να έχουν ακριβώς τα ίδια ωφέλη. Αν όλοι έχουν αποφασίσει ε, να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα πρέπει να γίνει και όχι να κολλήσουμε στο πώς αποκαλούμε την περιοχή ο καθένας μας. Ε, γιατί έτσι δεν υπηρετούμε την Ιρλανδία. Dziękujemy panie pośle. Poprawki do jutra do godziny 13. Przyjęcie projektu. Σας e- ευχαριστώ όλους. 22 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο θα ψηφίσουμε την ε, μεθεπόμενη Δευτέρα. Ίσως να ακούσουμε πάλι κάποιες επικρίσεις από τον ΤΕΣ και άλλους, αλλά σας παρακαλώ δείξτε κατανόηση. Επόμενη συνεδρίαση 8 Οκτωβρίου, 3 με, 10, με 6.30 ε, και το επόμενο πρωί στις 9 Οκτωβρίου και απόγευμα. Ολοκληρώσαμε πριν από τον χρόνο που είχε προβλεφθεί για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Κάποιες φορές ζητάμε κάποια λεπτάκια παραπάνω από τους Ζερμενείς, ενώ τώρα τελειώσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.